υπόψη τη νέα πραγματικότητα αυτή. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Αντοκίνε. Ε, τελείωσε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο ε, το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Μια μικρή ανακοίνωση πριν περάσουμε στην επόμενη συζήτηση. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι η κυρία Πασκάλ Γκρουνή αντικαθίστανται από τον κύριο Φιλίπ Μπουλόν από τις 15 Δεκεμβρίου 2010. Θέλω να καλωσορίσω τον νέο συνάδελφο. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στην αίθουσα. Όχι μάλλον αυτή τη στιγμή. Ε, Πάντω θα ακούσει το μήνυμά μου και με βάση το άρθρο 3 παράγραφο 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο βαθμό που οι αρμοδιότητέ του δεν έχουν επαληθευτεί, έχουν ή δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, ο κύριο Φιλίπ Μπούλα ε, θα εδρεύει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα όργανά του θα απολαμβάνει τα δικαιώματά του υπό τον όρο ότι έχει κάνει δήλωση ότι δεν ασκεί ε, κάποια σύμβατη λειτουργία ή ε, αξίωμα μαθή του, Ευρωπαϊκού, του Ευρωβουλευτή. Και τώρα πάμε στην έκθεση Αρλάκη για τη νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πίνο Αρλάκη, για τέσσερα λεπτά. Thank ε, Ευχαριστώ. Λέδι Άστον, συνάδελφοι, η έκθεση αυτή εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από την ΑΦΕΤ. Βασίζεται σε ε, εκτεταμένες διαβουλεύσεις στην Καμπούλ και στις Βρυξέλλες. Είναι μία απόπειρα να εξηγήσουμε ένα παράδοξο γιατί τόσα λίγα έχουν επιτευχθεί στο Αφγανιστάν παρά το γεγονός ότι συμμετέχουμε νέα χρόνια σε αυτή την περιοχή. Από το 2001 οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τύχησαν 300 δις ευρώ και αρκετές χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και 40 δις έχουν δαπανηθεί από πολιτικής πλευράς, δηλαδή 30 φορές το ΑΕΠ του Αφγανιστάν παρά τις ε, τεράστιες προσπάθειες το Αφγανιστάν είναι ο πρώτος παραγωγός ναρκωτικών. Είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο όπου για την πλειοψηφία του αφγανικού λαού η ζωή είναι πολύ μικρή και κακής ποιότητας όπως ήταν στην Ήπειρό μας 4 ή 5 αιώνες πριν μητρική εθνισμότητα είναι της τάξης των 20.000 ε, ετησίως. Η απάντηση σε αυτό το παράδοξο δεν είναι απλή. Το όπιο και η αντίσταση είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Είχαμε την αυταπάτη μιας μεγάλης και γρήγορης νίκης. Επίσης, η νομιμότητα της κεντρικής κυβέρνησης έχει υπερτιμηθεί καθώς και η αρρωγή για την βοήθεια αυτής της χώρας, η διεθνή αρρωγή. Η έκθεση αυτή δεν θέλει να απλουστεύσει το όλο ζήτημα. Δέχεται την πραγματικότητα ως έχει και θεωρούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε νέα προσέγγιση στην πολιτική μας. Εμείς βλέπουμε από ευρωπαϊκής πλευράς πώς έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη το θέμα από μια οπτική γωνία που δεν συμπεριλαμβάνει την ε, αμερικανική θεώρηση. Μας ενδιαφέρει το πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες βλέπουν το θέμα του Αφγανιστάν που δεν πιστεύουν σε μία στρατιωτική λύση. Επειδή 65 χρόνια πριν θεωρήσαμε ότι η εμπόλεμη κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Εμείς αποστρεφόμαστε τον πόλεμο και η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει αυτό το αίσθημα. Ως προς το ειδικό θέμα του Αφγανιστάν πιστεύουμε σε μια πολιτική προσέγγιση ως εναλλακτική από την χρήση της βίας. Η προσέγγιση μας δεν είναι αφελής. Δηλαδή δεν είμαστε υπέρ μιας Αφροδίτης και κατά ενός Άρη. Πιστεύουμε στην ανθρώπινη αλληλεγγύη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση όπως την Αφγανική που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το καρότο και το μαστίγιο. Προτείνουμε μία στρατηγική που δεν αποκλείει και κατασταλτικά μέσα. Η ασφάλεια είναι ύψης της σημασίας κατά της ε, τρομοκρατίας. Και το Κοινοβούλιο αυτό πιστεύει ότι οι ειρνευτικές δυνάμεις και η πολυμερής διπλωματία καθώς και οι εγχώριες διαπραγματεύσεις θα μειώσουν την φτώχεια. Θα φτάσουμε σε δημοκρατικά δημοκρατική διακυβέρνηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των, δικαιωμάτων με συγχωρείτε των γυναικών. Πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν πολύ σωστά από το σύστημά μας και θα ήθελα η κυρία Άστον να ε, συμμεριστεί την άποψη του Κοινοβουλίου στην προσπάθειά μας αυτή. Το λόγο έχει η ύπατη εκπρόσωπος για να αντιδράσει σε αυτή την ε, έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να μνημονεύσω τον Ρίτσαρτ Χόλπρουκ, αφοσιωμένο διπλωμάτη ε, και υπερασπιστή της ειρήνης και καλό μου φίλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρλάκη για την πλήρη έκθεσή του και την δουλειά που έχει κάνει, που ξέρω ότι έχει οδηγήσει σε μια πλούσια συζήτηση στο Κοινοβούλιο του τελευταίους μήνες. Εγώ προσωπικά προσλέπω στην συνεργασία μαζί του και άλλους συναδέρφους από το Κοινοβούλιο στους επόμενους μήνες, ε, κάτι που εγώ θεωρώ ότι αποτελεί κρίσιμη φάση στις σχέσεις μας με το Αφγανιστάν. Όπως είπε ο κύριος Αρλάκη, τα προβλήματα του Αφγανιστάν αφορούν όλους μας. Ο εξτρεμισμός, ε, τα ναρκωτικά ε, καταφτάνουν στη θέση, στους δρόμους της Ευρώπης. Θέλουμε να εμποδίσουμε το Αφγανιστάν ε, να γίνει ασφαλής λιμένας για τους τρομοκράτες ε, και εξτρεμιστές. Είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον ε, και, πιο, και μέλλον με ευμάρια για τους ανθρώπους του Αφγανιστάν. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μακροπρόθεσμα στο Αφγανιστάν. Έχουμε ένα πρόγραμμα βοήθειας μέχρι το 2013 και είμαι βέβαιη και μετά από αυτό. Έχουμε αυξήσει ε, την ε, βοήθειά μας από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την ε, κοινωνική ευημερία, την το κράτος ε, δικαίου, την υγεία κλπ. Έχω αναφέρει επανειλημμένα τον τομέα της υγείας. 8% του, της χώρας έχει κάποιο είδους πρόσβαση σε ε, πρωτογενή ε, υγειονομική περίθαλψη. Από τα στοιχεία του ΟΗΕ γνωρίζουμε ότι σε σχέση με το 2001 40.000 λιγότερα παιδιά μωρά πεθαίνουν κάθε χρόνο στο Αφγανιστάν. Αυτό ε, οφείλεται στην ε, καλύτερη προγεννητική περίθαλψη. Θέλουμε Συγγνώμη, το 50% της βοήθειάς μας περνάει είτε μέσω ε, εθνικών προγραμμάτων ή μέσω ε, ε, καταπιστευματικών οργανισμών και αυτό είναι πολύ καλό για να παγιωθεί η οικειοποίηση από τους Αφγανούς. Υπάρχει όμως ακόμα χώρος για βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά βλέποντα το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδιαίτερα με την άφηξη του Ουζάκα που έφτασε στο Αφγανιστάν τον Απρίλιο μέσω του σχεδίου δράσης για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν ε, που εγκρίθηκε πέρσι τον Οκτώβριο από το Συμβούλιο έχουμε βελτιώσει τις δράσεις μας. Το σχέδιο δράσης ε, συντονίζει τα μέσα που χρησιμοποιούμε και τα ευθυγραμμίζει με τι πολιτικέ προτεραιότητές μα, ιδιαίτερα αυτέ που προκύπτουν από τη διάσκεψη τη Καμπούλ, στην οποία συμμετείχα τον Ιούλιο. Η ευθυγράμμιση της ε, προσέγγισής μας αποτελεί στοιχείο κλειδί του σχεδίου μας. Η Ευρωπαϊκή η ε, ε, αρμόδιοι υπουργοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την Προεδρία μου συζήτησαν τα θέματα αυτά την προηγούμενη εβδομάδα στι Βρυξέλλε. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο με φέρνει στο μήνυμα κλειδί που έχω για σήμερα, ότι η εφαρμογή των ε, συστημικών στρατηγικών μας ε, πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Ε, το στρατηγικό πλαίσιο υπάρχει ήδη και στο στρατιωτικό και στον πολιτικό τομέα. Μαζί με τους δύο προέδρους συμμετείχα στην συνάντηση της ISAF στη Λισαβόνα την προηγούμενη μήνα όπου συμφωνήθηκε το μεταβατικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Ε, τρεις φορές συνάντησα τον ε, ε, στρατηγό τους τελευταίους μήνες ε, και πιστεύω ότι οι στρατηγίες πραγματικά αρχίζουν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική πλευρά. Ε, είχαμε μια επιτυχημένη διάσκεψη της Καμπούλη. Η αυγανική κυβέρνηση θα πρέπει να επενεθεί για ε, την διοργάνωση ε, της εκδήλωσης αυτής ε, τον Ιούλιο. Δεν ήταν η συνήθις επανάληψη ετοιμάτων και υποσχέσεων από χορηγούς το να διοχετεύουμε τις προσπάθειες μας σε εθνικά προγράμματα των ε, Αφγανών είναι ε, σημαντικό βήμα, διότι έτσι ε, μπορούμε να... Έτσι έχουμε ανοίξει τον δρόμο για την μετάβαση στην αφγανική οικειοποίηση σε διάφορους τομείς. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλή έξοδο του στρατού από το Αφγανιστάν χωρίς να ε, υπάρχει σταθερότητα. Ε, καλύτερους ε, θεσμούς, καλύτερη διακυβέρνηση, πρόσβαση σε κάποιες βασικές υπηρεσίες και το κράτος δικαίου είναι εξίσου σημαντικά με την στρατιωτική ασφάλεια. Θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν για να δημιουργήσουμε ε, ε, ε, αρμόδιους και υπεύθυνους θεσμούς, ιδιαίτερα στο υποεθνικό επίπεδο, στο περιφερειακό επίπεδο. Θα εργαστούμε ε, ώστε να οικοδομήσουμε ε, αφγανικούς ε, θεσμούς για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την διαφθορά. Και θα ήθελα να κλείσω με λίγα λόγια για κάποιες αυγανικές προσπάθειες. Οι δικές μας προσπάθειες θα πετύχουν μόνο ε, όταν ε, γίνει πιο ε, συμμετοχική η κυβέρνηση και έχει περισσότερη αίσθηση λογοδοσία. Αυτή τη στιγμή το μισό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας είναι περιθωριοποιημένο και βλέπουμε από άλλα μέρη του κόσμου ότι η συμμετοχή των γυναικών ε, ε, στις κυβερνητικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντικό. Ε, μου έκανε εντύπωση το δυναμικό αυτό το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο στη συνάντησή μου με γυναίκες πέρσι στο Αφγανιστάν η υποστήριξη γυναικών βουλευτών στο Αφγανικό Κοινοβούλιο ή ε, η ενθάρρυνση της συμμετοχής γυναικών σε τοπικά προγράμματα ε, είναι τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, ε, μέσω του προγράμματος που χρηματοδοτούμε μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα από το 2002. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Αρλάκη που τόνισε τόσο σημαντικά θέματα στην έκθεσή του. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η στιγμή που εμφανίζεται η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκέρεντσε. Από την Επιτροπή Ανάπτυξης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Αφγανιστάν δεν έχει πολλές επιλογές. Πρώτον, το status quo δεν είναι ρεαλιστική δυνατότητα, γιατί ε, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχουν ανακοινώσει η μία μετά την άλλη χώρα που συμμετέχουν, δηλαδή την αποχώρησή του και επομένω δεν εγγυώνται πια την ασφαλειά του. Η επιστροφή ε, στην κατάσταση πρώτου 2000 ούτε αυτή είναι επιλογή. Και τα δίκτυα των τρομοκρατών ε, θα, ε, θα μπορούσαν να έρθουν σε μια διελκυστίδα με, τις, με τους ξένους στρατιωτικές δυνάμεις. για το κατά πόσο μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με τους Ταλιμπάν, πώς μπορώ να μιλήσω. Ε, υπάρχουν εξάλλου μετροεπαθείς ε, Ταλιμπάν. Ε, ας ρωτήσουμε εξάλλου και τις γυναίκες ε, ε, που έχουν ζήσει ένα πραγματικό εφιάλτη και που τώρα μόλις βρήκα μια κάποια ελευθερία. Το θέμα είναι να ε, δρεωθούν τα κεκτημένα και να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία και ανάπτυξη. Ο Καρζάη θέλει να ενσαρκώσει αυτή την επιλογή, αλλά έχει ένα βασικό εμπόδιο, την προσωπικότητά του. Όσο δεν υπάρχει ε, αξιόπιστη ε, εναλλακτική λύση, είναι η μόνη επιλογή που έχουμε, ε, ο Καρζάη δηλαδή. Τώρα, από τις πολιτικές ομάδες, ο πρώτος είναι ο κύριος Κασουλίδης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βασική μας θέση σε αυτή την έκθεση είναι ότι μια στρατηγική κατά του Αντάρτικου ε, στο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ τον κύριο Αρλάκη που το κατανοεί αυτό. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει ε, όμως να έχει αρκετό χρόνο για να δώσει αποτελέσματα με βάση το χρονοδιάγραμμα του Πρόεδρου Ομπάμα. Ε, το 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πλήρη αυγανοποίηση των δυνάμεων του στρατού και της αστυνομίας. Φυσικά ε, η λύση είναι πολιτική με μια συμφωνία ε, που θα την πετύχουμε ε, με διαπραγματεύσεις με όλους τους, τις αφγανικές πλευρές. η σύγκρουση με τους Ταλιμπάν είναι αφγανική υπόθεση. Αλλά όμως μπορεί να γίνει η πρόοδος όταν οι αντάρτες σταματήσουν να είναι σε αυτή τη θέση ισχύω. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη βοήθεια που δίνουμε μέσω των αναδόχων, ούτως ώστε να υποφελεί το τοπικός πληθυσμός και χωρίς να πληρώνουμε λεφτά ε, για την προστασία ε, από τους αντάρτες ε, των διαδρομών που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τις προμήθειες. Είναι σημαντική η ασφάλεια για τις ανθρώπινες ζωές. Δεν μας αρέσει η παράγραφος 71 που καταδικάζει τη χρήση των ε, ελικοπτέρων που είναι ε, βασικό στοιχείο της στρατηγικής ε, καταπολέμησης του Αντάρτικου. Οι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί τι θα σκεφτούν αν εμείς καταδικάσουμε ένα τόσο σημαντικό όπλο κατά των ανταρτών. Θα ήθελα να καταψηφίσετε, συνάδελφοι, αυτή την, το τρίτο τμήμα της παραγράφου αυτής, της παραγράφου 51. Ο Νόιζερ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Λέδη Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια πολλών αποστολών ε, με βάση ε, αποφάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στο Αφγανιστάν. Πολλοί νέοι Ευρωπαίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αφγανιστάν, πολλοί έχουν ε, ε, τραυματιστεί σοβαρά ή ε, υποφέρουν από πράγματα που συνδέονται με τις στρατιωτικές προσπάθειες. Ε, χιλιάδες Ευρωπαίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε μέρα για να βοηθήσουν το Αφγανιστάν να έχει καλύτερο μέλλον. Όλοι εμείς έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε Πώ ε, μπορούν οι προσπάθειες της ε, Ευρώπης στο Αφγανιστάν να οδηγηθούν σε επιτυχές αποτέλεσμα και πόσο θα διαρκέσουν οι προσπάθειες εκεί. Τι θα πρέπει να αλλάξει, ποιοι είναι οι στόχοι της νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφγανιστάν. Χρειαζόμαστε βελτιωμένες ε, προσπάθειες για για πολιτική ανοικοδόμηση. Χρειαζόμαστε νέα κατάρτιση της αστυνομίας και του δικαστικού. Ε, ξέρουμε ότι δεν, μπορούμε να έχουμε στρατιωτική λύση και γι' αυτό οι προσπάθειες μας για πολιτική λύση ε, της ε, σύγκρουσης θα πρέπει να ενταθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινή εξωτερικής πολιτικής. Η αφγανική διαδικασία συμφιλίωσης με την συμμετοχή ε, μετριοπαθών ε, Ταλιμπάν θα πρέπει να ε, προωθηθεί. Συγκεκριμένες προσπάθειες, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν στόχο σταθεροποίηση της κατάστασης. Εδώ εμπίπτει και η καταπολέμηση της καλλιέργειας και του εμπορίου ναρκωτικών. Η στρατηγική μας περιέχει καλές προτάσεις από την αφγανική κυβέρνηση. Απαιτούμε ε, σαφή βούληση για καλύτερη, δηλαδή μη ε, διαφθαρμένη διακυβέρνηση. Η νέα στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο ε, εάν δεν παραμένει παθητική, αλλά ενεργά έχει ενεργή παρουσία και με συμμετοχή των γειτονικών μελών. Λέδη Άστον, σας στηρίζουμε απόλυτα. Ευχαριστώ lady ashton Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέδη Άστον, σας ευχαριστώ που αναφέρατε τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Ε, είναι σημαντικό να τον θυμόμαστε σήμερα που μιλάμε για το Αφγανιστάν. όλα τα κράτη του κόσμου έχουν πρόβλημα με το Αφγανιστάν. Ε, σήμερα διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση. Καθημερινά όμως βλέπουμε νέα θύματα ε, στρατιωτών ε, αλλά και πολιτών. Ε, έχουμε στην έκθεση του Πίνο Αρλάκη κάποιες αναλλακτικέ ε, προτάσεις. Ε, η έκθεση αυτή αναφέρει ε, πλεονεκτήματα και ελλείψεις των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σήμερα είναι σαφές ότι ε, το βασικό πρόβλημα δεν είναι η παρουσία της Αλκάιντα στο Αφγανιστάν. Το πρόβλημα ε, της τρομοκρατίας φαίνεται να έχει μεταφερθεί σε γειτονικές χώρες. Η έκθεση αναφέρει μακροπρόθεσμη λύση στο Αφγανιστάν όπου να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και παιδιών και γυναικών. Κάτι τέτοιο μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την στενή συνεργασία ε, και των, της αφγανικής κυβέρνησης, ε, της κοινωνίας ε, και των τοπικών ηγετών. Θα Πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να μπορεί να γίνει αποδεκτή και με βάση τις αξίες ε, του λαού του Αφγανιστάν. Ε, είναι πολύ σημαντικό σημαντική η έκθεση αυτή διότι ε, δείχνει τα προβλήματα που υπάρχουν στα Αφγανιστάν ε, και μας ε, ενθαρρύνει για την συνέχιση μιας υπεύθυνης πολιτικής στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Κύριε Νίλσον, ενάμιση λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρλάκη για την επικοδομητική ατμόσφαιρα με στην οποία εργαστήκαμε. Αυτή η έκθεση προτείνει μια τίμια και ακριβή ανάλυση των ελλείψεων της ε, διεθνούς κοινότητας ε, στο Αφγανιστάν το 2001 μέχρι τούδε. Ε, δεχόμαστε το βασικό μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική λύση, ο πόλεμος κοστίζει ακριβά, ε, κοστίζει ανθρώπινες ζωές ε, και σε επίπεδο αμάχου πληθυσμού αλλά και σε επίπεδο στρατιωτών. Ο πόλεμος ενδυναμώνει του Ταλιμπάν. Η μόνη λύση είναι πολιτική. Αυτό περιμένουν ε, οι Αφγανοί. Είναι να επενδύσουμε στην ανάπτυξη της χώρα τους, ε, στην καλή διακυβέρνηση, ε, στη δημιουργία ενός ε, δικαστικού συστήματος. Τα προβλήματα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίως των γυναικών είναι πάρα πολλά. Η πρόσφατη έκθεση το, της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν δείχνει την ανικανότητα της κυβέρνησης του Αφγανιστάν να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Όσο οι γυναίκες και τα κορίτσια, λέει, ε, υφίστανται πρακτικές που επιδεινώνει ή του στερεί τα δικαιώματά τους, δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικές, ε, ουσιαστικά βήματα προόδου στο Αφγανιστάν. Για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, χρειαζόμαστε όχι μόνο συνταγματικά και ε, δικαιώματα και δικαστικά δικαιώματα επί χάρτου, αλλά κυρίως την ε, γρήγορη και κατάλληλη εφαρμογή τους. Η Εθνική Συνέλευση έχει ελάχιστη επιρροή στη χώρα. Το βασικό στοιχείο της εξουσίας βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου Καρζάη. Εάν δεν είναι αργά, μια υποστήριξη για την ενδυνάμωση τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου θα πρέπει να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ του διάφορου φορεί και κυρίω στο κοινοβούλιο που μόλι εξελέγει. Ευχαριστώ κύριε Νίλσεν. Τώρα ο κύριος Στίβενσον για δύο λεπτά. Εκτός μικροφώνου. For the past year I've served την τελευταία χρονιά ήμουνα εκπρόσωπος ε, του Προεδρεύοντος ε, του ΟΣΑ ε, για το Καζακστάν ε, ε, Βαρόνι σας έχω στείλει ε, αντίγραφο της έκθεσής μου που αναφέρει τα προβλήματα της Κεντρικής Ασίας. Ένα από τα βασικά προβλήματα της Κεντρικής Ασίας είναι η διασυνοριακή χρήση του ύδατος. Όπως ξέρετε υπάρχει σημαντική τάση ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής Ασίας όσον αφορά την χρήση του ύδατος. Ε, ένα στοιχείο που ε, είδα, που νομίζω ότι έχει αγνοηθεί από πολλούς που λαμβάνουν αποφάσεις στη Δύση, είναι ότι η βάση της αυγανικής οικονομίας είναι η γεωργία. Και οποιαδήποτε ανοικοδόμηση ε, της οικονομίας του Αφγανιστάν θα συνεπάγεται ε, σημαντικές επενδύσεις στην ε, γεωργία ε, ώστε να αλλάξουν καλλιέργειες οι γεωργοί και αντί για όπιο να καλλιεργούν ροδιές. Αυτό σημαίνει ότι Αυτό όμως ε, απαιτεί ε, σημαντικές ποσότητες νερού, το οποίο σημαίνει ότι ε, οποιαδήποτε προσπάθειά μας να αλλάξουν καλλιέργειες στο Αφγανιστάν μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα με το νερό. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και τα αρδευτικά συστήματα και οποιαδήποτε προγράμματα ενέργειας με υδροηλεκτρικά εργοστάσια θα πρέπει να κατασκευαστούν πολύ προσεκτικά ώστε να μην οδηγήσουν σε προβλήματα ε, χωρών ε, πιο κάτω στα ίδια ποτάμια. Ε, ευχαριστώ ο κύριος Higgins για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ο πόλεμο ε, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών ε, στο Αφγανιστάν είναι καταστροφή για τον αφγανικό λαό. 40.000 υπολογίστε ότι σκοτώθηκαν πέρσι. Είναι καταστροφή και για του νέου ε, ανθρώπου του Αφγανιστάν που αναγκάζεται να παλέψουν, να αγωνιστούν στο στρατό, στους στρατούς του ΝΑΤΟ και του Αφγανιστάν. Ίσως 500 από αυτούς να πέθαναν πέρσι. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι ζωφερή. Πολλοί άνθρωποι ο αριθμός ε, όσων ζουν ε, στη φτώχεια έχει αυξηθεί ε, και υπάρχει και ένα σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο το ότι τρισεκατομμύρια δολαρίων έχουν σπαταληθεί για πολεμικό εξοπλισμό. Ο πόλεμο στο Αφγανιστάν ξεκίνησε όχι για να προωθηθούν τα συμφέροντα του ε, αφγανικού λαού, αλλά για να προωθηθούν τα οικονομικά συμφέροντα της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και θα πρέπει από τους διεφθαρμένου πολέμαρχου και τον Καρζάη να πάρουμε την εξουσία και να την δώσουμε στα χέρια των γεωργών, των φτωχών που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν του όρους αυτούς προς όφελος του λαού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλτερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ως ε, εισηγητής για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι, έναντι του Ιράν θα ήθελα να πω ότι ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτό το ψήφισμα υπέρ του Αφγανιστάν και αυτό που με ενδιαφέρει είναι η επιρροή του Ιράν στο Αφγανιστάν της Ισλαμικής αυτής δημοκρατίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει την επιρροή του Ιράν στο Αφγανιστάν και ποιες είναι οι συνέπειες. Θα ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις και φαντάζομαι ότι η ύπατη εκπρόσωπος μάλλον θα μου απαντήσει γραπτός για να μου απαντήσει διεξόδικα. Μιλώ για τις απελάσεις προσφύγων Αφγανών από το Ιράν. Αυτό έχει χαρακτήρα αποσταθεροποίησης στη χώρα. Επίσης, συμμερίζεστε την ανάλυση της αφγανικής κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία μπαίνουν τρομοκράτες στην αφγανική γη μέσω αυτών των προσφύγων. Επίσης, τι θα κάνετε έτσι ώστε η Τεχεράνη να μην χρησιμοποιεί αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία για να πιέζει πολιτικά την Καμπούλ. Ο κύριος Γκρίφιν για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, αυτή η έκθεση στην ουσία οδηγεί στην ε, κατάρρευση της ε, Βρετανικής θέσης για τον Αφγανικό πόλεμο. Δεν ξέρω ε, ποια ακριβώς είναι τα θύματα, ξέρω όμως πώς στάθηκε η Βρετανία, τι θέση ακολούθησε η Βρετανία σε αυτό το θέμα. 18 άτομα έχασαν τη ζωή τους από το Λίβερπουλ, από το Λάνκασαρ, από το Σέλιμπριζ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 lance corporal jordan bancroft burnley kingsman darren deedy bolton guardsman christopher davis st helens. What a criminal... Αυτός ήταν ο κατάλογος των θυμάτων των Βρετανών στρατιωτικών. Δυστυχώς χάθηκαν πολλές ζωές, αλλά δεν ε, μας λέει η Βρετανία γιατί ή γιατί δεν πρέπει να ε, πολεμά. Το Westminster είναι αυτό που αποφασίζει αν θα πρέπει να πολεμήσουμε ή να μην πολεμήσουμε. Και κάποια στιγμή πρέπει ο Μπλερ ε, και ο Κάμερον να μπουν στο, να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει. Ο κύριος Μάουρο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα τεράστια προβλήματα που παραμένουν στο Αφγανιστάν ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση μια νέα λογική. Δηλαδή, με νέο καθορισμό των προτεραιοτήτων σε σχέση με τις μέχρι τούδε προτεραιότητες. Συμφωνώ επίσης το γεγονός ότι ο πρόεδρος Καρτζάη έχει θέσει ως στόχο το 2014 ως έναρξη της περίοδου όπου μόνο οι, δυνάμεις, οι αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας θα, θα πάρουν τον έλεγχο ε, για τις διάφορες επαρχίες για το θέμα της ασφάλειας. Όλα αυτά όμως δεν πρέπει να σημαίνουν ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το Αφγανιστάν εμείς ως διεθνής κοινότητα. Η συνεργασία με το Αφγανιστάν θα πρέπει να ενδυναμωθεί αντίθετα ε, από όλες τις πλευρές. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις στην οικονομία, γιατί αυτό σημαίνει επενδύουμε πραγματικά στη σταθερότητα της χώρας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Δηλαδή να έχουμε ένα μοντέλο συνεργασίας που θα βασίζεται στον διάλογο που συμπεριλαμβάνονται όλοι, ε, οι τοπικοί φορείς, ε, η κοινωνική πραγματικότητα κτλ. Αλλά όπως σωστά λέει και η έκθεση, δεν μπορεί να υπάρξει ε, σταθερότητα χωρίς να εγγυάται το κράτος στην ασφάλεια των πολιτών του και να αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Με αυτή την έννοια, καλώ τον εισηγητή να ξαναδεί αν μπορεί, μέσω μιας τροπολογίας προφορικής ίσως, το τμήμα για την χρήση των τηλεκατευθυνόμενων αεροπλάνων ε, σε διάφορες επιχειρήσεις ε, στο Αφγανιστάν. Δηλαδή άλλο είναι να πούμε ότι απαγορεύονται αυτά τα αεροπλάνα, άλλο είναι να λέμε ε, να περιορίσουμε τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για να μην πλήξουμε ας πούμε τον άμαχο πληθυσμό. Νομίζω ότι ο εισηγητής ε, έχει την ευαισθησία για να καταλάβει ε, πώς μπορούμε να, αναδιατυπώσουμε αυτό το σημείο και εμείς θα τον υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο. Ο κύριος Βίγγενιν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Σήμερα συζητάμε για ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του 2010 σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Θέλω να υποφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση. Τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας σημαίνει ε, μας μιλούν για μεγαλύτερη παιδική θνησιμότητα, μεγαλύτερο αναλφαβητισμό, ε, χειρότερη υγεία. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Μία εβδομάδα στρατιωτικών δαπανών ε, κοστίζει όσο θα κόστιζαν έξι σχολεία. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι πολύ πλήρη, αλλά αυτά διαθέτουμε τώρα. Από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ξόδεψαν πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς αποτέλεσμα για αυτή τη χώρα η επιλογή για την εκπαίδευση των Αφγανών αστυνομικών δεν καλύπτει τα στοιχειώδη κριτήρια. Το 1 πέμπτο αυτών είναι ναρκωμανείς και οι υπόλοιποι είναι αναλφάβητοι. Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε μια νέα στρατηγική, αλλά επίγνωση του προβλήματος. Η μόνη λύση είναι η πολιτική λύση. Να συμμετάσχουν οι φορείς, ε, να συμμετάσχουν οι πολίτες, να βρούμε μια μακροπρόθεσμη λύση και να σταματήσει η παραγωγή των ναρκωτικών. Χάγκλουντ, δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Αρλάκη για την πολύ καλή δουλειά που έκανε πάνω στην στρατηγική αυτή. Αυτό μας δείχνει και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε, μας δείχνει και τα λάθη που έχουν γίνει. Ελπίζω να μπορούμε να εξάγουμε καλά συμπεράσματα όσον αφορά το τι έχουμε να μάθουμε και το τι πρέπει να κάνουμε στο Αφγανιστάν. Υπάρχει μια ριζοσπαστική αλλά σημαντική ε, σκέψη σχετικά με το αν θα πρέπει να έχουμε συζητήσεις με τους μετριοπαθείς Ταλιμπάν. Αυτός μάλλον είναι ο μόνος τρόπος προόδου, αν και είναι δύσκολο να ορίσει κανείς τι είναι ο ε, μετριοπαθής Ταλιμπάν. Ε, δεν είναι πολύ σαφής ε, ο όρος αυτός ακόμα στα μυαλά μας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι τα χρήματα βοήθειας που δίνονται στο Αφγανιστάν και το τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Αφγανούς στο μέλλον. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και τους εκλογείς μας στις χώρες μας, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την κατάχρηση των πόρων που δίδονται στο Αφγανιστάν. Ο ρόλος του Πακιστάν είναι κρίσιμος. Η διεθνής κοινότητα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο ε, στο να ασκήσει πίεση στο Πακιστάν. Όσον αφορά τη δική μου χώρα, η συζήτηση αυτή τη στιγμή αφορά αποκλειστικά το αν θα υπάρχει παρουσία φιλανδικών στρατευμάτων, πού θα βρίσκονται αυτά κλπ και στη Σουηδία είδαμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Τσαρνέκη. Ευχαριστώ. Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουν παρατηρητής στις αυτόνομες παλαιστινιακές ε, περιοχές στην Παλαιστινιακή περιοχή δηλαδή, και θυμάμαι ότι κάποιος εκπρόσωπος μου είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι της Χαμάς είναι καλοί, πολιτισμένοι, ίσως καλό θα ήταν να διαπραγματευτούμε μαζί μας, μαζί τους. Ε, σήμερα έχω την αίσθηση ότι τα έχω ξανακούσει όλα αυτά. Ε, πάλι τα ίδια ακούω. Ακούμε ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε, λέει, με τους μετριοπαθείς Ταλιμπάν. Μα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει αυτό το πράγμα είναι μια έννοια σαφώς προσδιορισμένη. Προσοχή. Κάνω έκκληση να δείξουμε προσοχή. Είναι αλήθεια ότι πολλοί στρατιώτες πέθαναν στο Αφγανιστάν ε, και πολλοί Πολωνοί στρα, ε, στρατιώτες πέθαναν εξάλλου και ότι ο πόλεμος ε, είναι δαπανηρός. η στρατηγική του ΝΑΤΟ επίσης είναι διφορούμενη. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο κύριος Ζουβά για δύο λεπτά. Ο Ζουβά. Κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι ο Σαρλάκη γνωρίζει καλά το Αφγανιστάν. Ε, από εμά είναι ένας από αυτούς που γνωρίζει καλύτερα αυτή τη χώρα και αυτή την περίπλοκη περιοχή. Αλλά ας πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Αυτό το κείμενο έτσι όπως έχει δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν συμφωνώ με το σύνολο των συναδέλφων που χαίρονται για το κείμενο αυτό και θα σα εξηγήσω γιατί. Νομίζω ότι αυτό το κείμενο καταρχάς ε, θέλει οπωσδήποτε εμείς οι Δυτικοί να είμαστε υπεύθυνοι για τα δεινά του Αφγανιστάν. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Καταρχάς, ο κ. Σαρλάκη γράφει ότι οι υγειονομικές συνθήκες ε, επιδεινώθηκαν από τη στιγμή που φτάσαμε εμείς εκεί. Κατά τύχη. Η κυρία Άστο μας είπε ακριβώ το αντίθετο. Κανένας δεν το παρατήρησε όμως αυτό. Δεύτερον, ε, στο εκτιμώντας Β, διαβάστε το. Ε, συνάδελφοι, οι δυτικέ ε, δυνάμει εμφανίζονται ω δυνάμει κατοχή. Τα κράτη-μέλη ε, τη συνέλευση αυτή που γνώρισαν κατοχή θα καταλάβουν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Τρίτον, στην παράγραφο 71 για, τους, για τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα. Εγώ ήμουν αξιωματούχο στο Αφγανιστάν, αξιωματικό στο Αφγανιστάν ω στρατιωτικό γιατρό. Και είδα ασθενεί ε, και Ταλιμπάν και Αφγανούς αλλά και ξένου και Ευρωπαίου. Ε, αν σήμερα πείτε στους ε, στρατιωτικούς μας δεν μπορεί να χρησιμοποιείτε αυτά τα αεροπλάνα, ε, σημαίνει ότι τους λέτε πάρτε ρίσκα. Εσείς να έρθετε σε επαφή με τους, ε, με τους Αφγανούς. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή και υπεύθυνη στάση των πολιτικών να λέμε τέτοιο πράγμα. Ε, ξέρω ότι ο πόλεμο είναι σκληρό και αδυσόπιτο, αλλά αυτόν τον αντιμιλιταρισμό θα πρέπει να τον σταματήσουμε. Αυτόν τον πρωτογενή αντιαμερικανισμό να το σταματήσουμε. Αυτό το αυτομαστίγωμα των δυτικών να το σταματήσουμε. Δεν είμαστε εμεί τα δεινά των Αφγανών. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Οι εχθροί είναι οι Ταλιμπάν, δεν είναι οι Αμερικάνοι ε, και δεν είναι οι δυτικέ δυνάμει, οι εχθροί. Όλα αυτά είναι περίπλοκα. Αλλά προσοχή, για τον προσοχή προς τον τρόπο που παρουσιάζουμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Σουβά. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπέρμαν. Για ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δέχομαι κυρία Άστον το ότι αποτίσατε φόρο τιμή στον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Τον είχα συναντήσει στο Ντέιτον και στις Βρυξέλλες και γνωρίζω τις ικανότητές του αλλά νομίζω ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να γνωρίσουν επιτυχίες στο Αφγανιστάν. Μιλάμε για 20.000 στρατιωτικές ε, δυνάμεις το 2001, 150.000 σήμερα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδώσει αυτή η στρατηγική. Μας ενδιαφέρει η ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας. Μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση, η υγεία. Θα πρέπει να ζήσουμε χωρίς όπιο. Θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές καλλιέργειες. Ακούμε ευσεβείς πόθους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά τίποτα δεν γίνεται ως προς αυτό. Και αυτό οδηγεί στην γενικότερη καταστολή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, ε, τη διοίκηση στο Αφγανιστάν. Ο κύριος Ζιόμπρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα αρρωγής στο Αφγανιστάν χωρίς εσωτερική σταθερότητα σε αυτή τη χώρα το, ο βασικός πυλώνας πρέπει να είναι η ασφάλεια και η καταστολή των εξεγέρσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ και με τη UPOL. Επίσης θα πρέπει να καταστήλουμε στο Πεσαβάρ τις δυνάμεις των Ταλιμπάν. Κατά το δυνατόν βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων προέρχεται από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους καλλιεργητές να μην καλλιεργούν όπιο, αλλά να προβούν σε εναλλακτικέ καλλιέργειες. Όπως είπε ο στρατηγός Πετρέους, ε, τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να επηρεάσουν την ε, κατάσταση της περιφέρειας. Ευχαριστώ, η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η υπόθεση της κατάστασης στο Αφγανιστάν παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη διεθνή κοινότητα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν εκεί στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά γιατί εκεί αναπτύσσονται και θα αναπτύσσονται στο μέλλον δυνάμεις που θα συνιστούν τρομοκρατικές επιθέσεις και θα δημιουργούν προβλήματα στη διεθνή κοινότητα. Ε, η αλήθεια είναι και πρέπει να το παραδεχθούμε ότι στο αφγανιστάν από τον 14ο αιώνα ακόμα υπήρχαν δυνάμεις αυτού του τύπου φονταμενταλιστικές και τρομοκρατικές. Πριν από 24 χρόνια, κυρία Άστον, το κοινοβούλιο μας ψηφίζοντας την έκθεση της Επιτροπής Έρευνας για τα Ναρκωτικά αφιέρωσε ιδιαίτερες σελίδες στο Αφγανιστάν με προβλέψεις για τη σημερινή κατάσταση που δυστυχώς βγήκαν αληθινές το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν μπορεί να κατασταλεί με καλλιέργειες ε, κυρία Άστον. Το πρόγραμμα καλλιεργιών των ΗΠΑ στην πραγματικότητα έχει αποτύχει. Το όπιο του Αφγανιστάν, το οποίο θεωρείται και το καλύτερο σύμφωνα με τους ειδικού όπως αναφέρουν, ε, ακριβώς χρηματοδοτεί όλες τις δραστηριότητες και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν και αλλού. Επομένως χρειάζεται και καταστολή αλλά κυρίως χρειάζεται αυτό που είπατε εσείς ίδια δηλαδή η προσπάθεια η αναπτυξιακή η προσπάθεια στον τομέα της υγείας στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας δηλαδή να υποδειχθεί στους ανθρώπους αυτούς ένα μοντέλο που θα το αγαπήσουν θα το συμπαθήσουν και θα το θέλουν για την ποιότητά τους στην ε, ζωή τους εν συνεχεία για να μπορέσουν να το ενσωματώσουν στην αντίληψή τους. και φυσικά ένα τέτοιο μοντέλο θα βοηθήσει τις γυναίκες γιατί πρόκειται περί μνημειώδους ε, υπόθεσης ε, δηλαδή η κατάσταση στην οποία μετέβαλαν τις γυναίκες οι ταλιμπάν. ήδη στις μουσουλμανικές χώρες οι γυναίκες βρίσκονται υπό φοβερή κατάσταση και φοβερή καταπίεση εκεί τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Ε, είναι ανάγκη η ευρωπαϊκή ένωση να παραμείνει ε, βαρόνια και οι παρεμβάσεις σας να είναι συνεχείς και να παραμείνει με το ευρωπαϊκό της πρόσωπο αυτό ακριβώς που αναφέρατε και εσείς οι ίδια. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Γιαννάκου. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ο θα πρέπει να τιμήσουμε τον ε, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, ο οποίος είπε πριν πεθάνει πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι αποφασιστική σημασίας για την ευρωπαϊκή και την ε, παγκόσμια ειρήνη και όπως είπε και ο Πίνο Αρλάκη θα πρέπει να περισσώσουμε την κατάσταση επανορθώνοντας τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν και προβάλλοντας αρρωγή προς τον αφγανικό λαό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγξουμε και τις ξένες δυνάμεις στην περιοχή αυτή. Βεβαίω το κράτος δικαίου δεν μπορεί να συσταθεί από διεφθαρμένους πολιτικούς. Όμως θα πρέπει να ελέγξει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση την κατάσταση έναντι των στρατιωτικών και σε αυτό θα πρέπει να συνεισφέρει και το Πακιστάν. Δεν θα πρέπει να προβάλλουμε μια πολιτική στρουθοκαλιμιλισμού. Πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια της ΙΣΑΦ και του ΝΑΤΟ μπορούμε να βοηθήσουμε την κατάσταση και να αντιμετωπίσουμε και το Πακιστάν παράλληλα. Ο κύριος Φιντάντσα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Ε, χαίρομαι και εγώ για την αποτίμηση φορού τιμή στο Ρίτσαρτ Χόλμπρουκ. Ε, αν είχατε δώσει αυτή την έκθεση στη δική μου πολιτική ομάδα, θα είχαμε ακολουθήσει τελείω τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του Αρλάκη. Ε, σήμερα, χάρη στις πολλές τροπολογίες από τη δική μας πολιτική ομάδα, νομίζω ότι η έκθεση είναι λιγότερο ιδεολογικά χρωματισμένη και αναγνωρίζουμε τα θετικά που έχουμε κάνει αυτά τα εννέα χρόνια, αλλά και τα προβλήματα. Και χαράσουμε ένα δρόμο, ε, ώστε να μπορέσουν οι αφγανικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σίγουρα η στρατιωτική λύση από μόνη της δεν αρκεί, αλλά θα πρέπει να ξαναπούμε ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες. Παραδείγματος χάρη, ε, κοντά στο Κανταχάρ, και επίσης έχουμε μεγάλες επιτυχίες εναντίον των ε, ανταρτών. Αυτό όμως ε, είναι εκ των όνου κάνευ αν θέλουμε να φέρουμε τους Ταλιμπάν ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ε, χάρη στη θυσία της ζωής πολλών νεαρών στρατιωτών του Ίζαφ, πολύ και από τη δική μου χώρα, το καταφέραμε αυτό. Ε, η όλη προσπάθεια δεν είναι μόνο στρατιωτική, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ε, χτίζουμε γε, ε, γεφύρια, σχολεία, έργα διάφορα που βοηθάνε την ανοικοδόμηση της χώρας. Υπάρχουν κάποια επίμαχα σημεία στην έκθεση, κυρίως αυτό που αφορά τη χρήση των ανεπάνδρωτων αεροπλάνων. Νομίζω ότι θα ήταν άκρητο να στερηθούμε το πολύ χρήσιμο αυτό εργαλείο, το οποίο ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο ειδικά σε περιοχές ε, στα βόρεια ανατολικά, που είναι πολύ δύσκολο να νικήσουμε εκεί χωρίς αυτό το εργαλείο του Ταλιμπάν. Ε, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό το σημείο, αλλιώς θα καταψηφίσω, αν δεν περάσει αυτό το σημείο, θα καταψηφίσω, όπως και η υπόλοιπη ομάδα μου, το, σημείο αυτό. Ο κύριος Στάλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Λέδη Άστον, συγχαίρω τον συνάδελφο Αρλάκη για την τολμηρή του έκθεση. Με, ε, ε, πολύ σωστά σήμερα μνημονεύουμε τον Ρίτσαρτ Χόλπρουκ και την συμβολή του στον αγώνα αυτόν. Θα ήθελα να αναφέρω ότι 1,6 δισεκατομμύρια ε, ε, ευρώ έχουν χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα αυτό. Ε, και ο πόλεμος ε, αυτός ε, έχει παρουσιάσει πολλά προβλήματα. Δεν έχω το χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες, ε, αλλά οι πολίτες μας περιμένουν από μας να δώσουμε τέλος στον πόλεμο αυτό. Ο πόλεμος αυτός έχει στοιχήσει πολλές ζωές και πολλά χρήματα. Έχει έρθει η ώρα να ε, φτάσουμε σιγά σιγά στην ειρήνη. Αυτό περιμένουν οι πολίτες μας, περιμένουν ε, πολιτική λύση, δεν πιστεύουν σε μια στρατιωτική ε, λύση. Κυρία Πασέσκου για δύο λεπτά. Χαίρομαι, διότι στα πλαίσια της ΑΦΕΤ οι πολιτικές ομάδες φτάσανε σε μία συμφωνία ως προς το, την έκθεση. Το κείμενο είναι πολύ πιο πιστικό από το προγενέστερα η κατάσταση στο Αφγανιστάν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρεύουμε διεθνώς. Οι οικονομικοί δείκτες δεν έχουν βελτιωθεί και πολύ συχνά έχουν ληφθεί αποφάσεις χωρίς να συμμετάσχουν οι αφγανικές αρχές. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που λείπει δεν είναι η πλαισίωση και οι μηχανισμοί. Χρειαζόμαστε μία στρατηγική προβολή σε σχέση με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταβάλει διεθνώς ε, μία προσπάθεια για να αντιμετωπίσει το Αφγανιστάν ως ένα κυρίαρχο ε, κράτος και θα πρέπει να βρεθεί μια πολιτική και διπλωματική λύση και όχι στρατιωτική. Γι' αυτό πιστεύω ότι μία από τις θέσεις κλειδί είναι να υποστηρίξουμε τη στρατηγική μας για να καταπολεμήσουμε τους εξεγερθέντες. Η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ της Λισαβόνας τόνισε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αφγανικές δυνάμεις μέχρι το 2014. Η χώρα μου δεν θα αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις έως ότου είναι το έδαφος του Αφγανιστάν ασφαλές για μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάσταση άρχισε από την ύπαρξη σοβιετικών δυνάμεων εκεί. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της ΙΣΑΦ θα πρέπει να επανατοποθετηθούν εκεί όπου υπάρχει ασφάλεια και όχι επισφάλεια. Εμείς θεωρούμε ότι η περιφέρεια αυτή θα παραμείνει ανασφαλής παρά το γεγονός ότι δρούν οι δυνάμεις ΙΣΑΦ επί του παρόντος. Το ρόλο θα πάρει τώρα ο κύριος Πρέντα για δύο λεπτά επίσης. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι δέχομαι αυτά που είπε ο κύριος Ζουβέ και θα ήθελα Καταρχήν να πω ότι λυπάμαι διότι ο τίτλος της έκθεσης δεν αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε εξ ονόματος της παγκόσμιας ε, κοινότητας, αλλά εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω υποβάλει τροπολογίες προς αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την συνεργασία με τους συμμάχους και όπως είπε ο συνάδελφος Ζουβέν με τις ΗΠΑ δεν χρειάζεται μία αποκλειστική και νέα στρατηγική. Θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα τη στρατηγική της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι εδώ και δύο χρόνια. Αυτή ήταν η στρατηγική και δεν χρειάζεται μια νέα οπτική γωνία. Επίσης θα πρέπει να μάθουμε από τα σφάλματα του παρελθόντος, τις συμμαχίες δηλαδή αλλά δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πριν την επέμβαση ήταν ιδεατή η κατάσταση. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Θα πρέπει να εξαφανιστούν οι Ταλιμπάν από αυτή την περιοχή και αυτός είναι ο μείζων στόχος μας στο Αφγανιστάν. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα θετικά στοιχεία της παρέμβασης και ιδιαίτερα ως προς το σχέδιο Πετρέους διότι στο Αφγανιστάν οι γυναίκες δεν έχουν δικαιώματα, πολύ λίγα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και πολύ, λίγοι, πολύ λίγες οδικές αρτηρίες υπάρχουν. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εξάλληψης της φτώχειας και των αναπτυξιακών στόχων έχουν μεγάλη σημασία για τη διασφάλιση της ειρήνης στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για μια πραγματιστική θεώρηση όπως αυτή της δικής μου ομάδας. Μην ξεχνάτε ότι έχουν υποβληθεί 400 τροπολογίες στην έκθεση Αρλάκη. Τώρα είμαστε στη διαδικασία Catch θα πάρουν το λόγο έξι συνάδελφοι. Είναι το περισσότερο που μπορώ να κάνω γιατί έχουμε καθυστερήσει τη συζήτηση. Ε, σας παρακαλώ για ένα λεπτό μόνο καθένας για να μπορούν να μιλήσουν και οι έξι. Από διάφορες πολιτικές ομάδες είναι αυτοί οι συνάδελφοι. Ε, ο κύριος Κολινό πρώτος έχει το λόγο. Δεν φαίνεται στην αίθουσα ο κύριος Κολινό. Λοιπόν, προχωρούμε. Ε, το λόγο κυρία Ντεσαρνέζ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θέλω να σας πω τα εξής. Αντίθετα από αυτό που υπόθηκε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη δική της στρατηγική για το Αφγανιστάν. Έχουμε στρατιώτες, άντρες, ε, οι οποίοι ε, δραστηριοποιούνται, έχουμε μέσα τα οποία έχουμε αναπτύξει στην περιοχή, πρέπει να έχουμε και το δικό μας προβληματισμό και τη δική μας στρατηγική. Δεύτερον, θα πρέπει τα χρήματα της διεθνούς κοινότητας να πάνε και στους Αφγανούς. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια. Κάθε μέρα το διαπιστώνουμε αυτό. Νομίζω ότι εν μέρη είναι και ευθύνη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ανθρωπιστικών οργανώσεων, αλλά σε μεγάλο βαθμό και η έκθεση δεν τονίζει αρκετά, ε, μεγάλο πρόβλημα ε, της κυβερνητικής διαφθοράς. Μια κυβέρνηση που είναι διεφθαρμένη, που δεν είναι δίκαια, δεν είναι αποτελεσματική. Τρίτον, το θέμα του πολιτικού διαλόγου. Έχει τεθεί. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κάνουμε διάλογο με τους Ταλιμπάν. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο. Γιατί το να κάνουμε ε, διάλογο ενώ είμαστε ε, σε θέση αδυναμίας ε, επιτόπου και ενώ έχουμε μιλήσει για αποχώρηση των τετικών δυνάμεων, θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να προβούμε σε πολιτικό διάλογο. Πολύνο είναι στην αίθουσα. Έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χάρη στι διάφορες τροπολογίες ε, συμφωνούμε με την έκθεση Αρλάκη και με τι προτεραιότητε που έχουν ε, αναφερθεί στην ε, έκθεση για την ανάπτυξη του Αφγανιστάν. Καταρχάς ένα καθιστός ε, διαφάνειας, την κατάρτιση της, των αστυνομικών δυνάμεων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και μια σοβαρή στρατιωτική και πολιτική στρατηγική. Είναι σημαντικό να τονίσουμε την εξασφάλιση του ελέγχου και της σταθεροποίηση της περιοχής, ούτως ώστε να αποδυναμωθούν οι Ταλιμπάν και η δράση τους. Ε, αυτό χάρη στην ειρηνευτική δραστηριότητα. Ε, πιστεύω ότι χάρη στην ε, συνεισφορά του ΕΛΚΕ το κείμενο είναι ισορροπημένο και τέλος θα ήθελα να αποτύσω φόρο τιμής στην, στη θυσία και στην απώλεια ζωής των στρατιωτών της πολυεθνικής δύναμης ΙΖΑΦ για την υπεράσπιση του τοπικού πληθυσμού. Νεβεντάλοβα έχει το λόγο τώρα παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι κανένας πόλεμος δεν φέρνει την ευημερία. Κάποιοι συνάδελφοί μας προβληματίζονται σχετικά με το αν πρέπει να υποστηρίξουμε κάποιο είδος αεροπλάνων ή όχι. Ε, εγώ δεν ε, θέλω να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες, θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Αρλάκη, την κατάσταση γυναικών και παιδιών στη χώρα αυτή θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Πολλά παιδιά στο Αφγανιστάν δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο και ε, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εάν δεν υποστηρίξουμε το ε, εκπαιδευτικό σύστημα, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνς θα πάρει το λόγο τώρα. Η έκθεση του κυρίου Αρλάκη βασίζεται σε σωστέ έρευνε και είναι πολύ ενημερωτική. Ε, επίκριση από πλευρά μου είναι ότι ε, θεωρεί ότι το Αφγανιστάν ε, δεν είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Μέχρι στιγμή έχουν σκοτωθεί 346 Βρετανοί στρατιώτε στο Αφγανιστάν, χιλιάδε άλλοι στρατιώτε καθώ και πολλοί πολίτες του Αφγανιστάν. Έχει ε, πέσει το προσδόκιμο ζωής. Ε, μας λέει ότι το 2001 δεν καλλιεργούνταν παπαρούνες στο Αφγανιστάν, ενώ μετά ε, από εννέα χρόνια συγκρούσεων το Αφγανιστάν παρέχει περισσότερο από το 90% της ηρωίνης στην Ευρώπη το ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών είναι μάλλον είναι σχεδόν παραπανεντικό δηλαδή δεν αντιστοιχεί στην ολόκληρη προοπτική θα πρέπει να δώσουμε τέλος στην κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Νικολάη έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και τα παιδιά και οι γυναίκες είναι ένα σημαντικό θέμα της έκθεσης Αρλάκη και Μιλάμε για, μιλάει για την νομιμότητα της στρατιωτικής παρέμβασης στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει να μιλήσουμε όμως για την αποδοτικότητα αυτής της επέμβασης, διότι πέρα από τους αισθηματισμούς διαρκεί 10 χρόνια αυτή η επέμβαση και δεν ξέρουμε κατά πόσο ε, είναι πραγματικά συνεπής και αποτελεσματική. Εμείς όλοι φέρουμε και θα πρέπει να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση αυτής της έκθεσης διότι μιλά για θέματα τα οποία συνήθως αποφεύγουμε και νομίζω ότι είναι μια έκθεση η οποία ε, μας δείχνει ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση για να δούμε πού έχουμε σφάλει και πού όχι. Αυτή είναι η δημοκρατία και η ευθύνη που φέρουμε. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. E, Κυρία Πρόεδρε, λέει Άστον, από τις εμπειρίες μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απ' έξω μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια μόνο αν το ζητάει αυτό ο λαός μετά από χρόνια στο Αφγανιστάν ε, ο λαός δεν καταλαβαίνει την επέμβασή μας. Ε, ε, στη χώρα μου λέμε ότι αν κάποιος δεν μπορεί να συμβουλεύσει δεν μπορεί να βοηθήσει και κανέναν. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορούν να δεχτούν βοήθεια οι Αφγανοί αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την βία κατά την παροχή βοήθειας. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς μπορούμε να παράσχουμε την βοήθεια ώστε να γίνει αποδεχτή από τον ε, λαό του Αφγανιστάν τους τοπικούς ε, πολιτικούς, ε, στους τοπικούς πολιτικούς θα πρέπει να δώσουμε ε, να, να παραδώσουμε την διοίκηση και ίσως τότε να είναι διατεθειμένοι να δεχτούν τη βοήθειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Πάσκου. Ο κύριος Πάσκου είναι στη yes για να υπάρχει ένα ευνομούμενο Αφγανιστάν που θα εμποδίζει την επανηθίδρυση του, της τρομοκρατίας είναι ένα στόχος του ΝΑΤΟ. Ο στόχος μας είναι μακρόπνος. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις προκλήσεις γι' αυτό. Πρώτον, ότι η βοήθεια που δίνουμε στο Αφγανιστάν δεν εντάσσεται στην παράδοση του Αφγανιστάν. Οι Αφγανοί, θα πρέπει να προσαρμοστούν, αλλά και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα πρέπει δηλαδή να συνδυαστεί ε, ε, η κατάσταση, οι μοντέρνες προϋποθέσεις με την παράδοση του Αφγανιστάν. Ε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει με τη στρατιωτική μας εμπλοκή μετά το 2014 θα αναλάβουν οι Αφγανοί τις ευθύνες τους. Τέλος, η τρίτη πρόκληση. Ε, το κοινό μας δεν θα έχει πια ευθύν, ε, υπομονή και θα μας αναγκάσει να επιταχύνουμε την αποχώρησή μας. Ε, θα, θα πούμε ε, νικήσαμε και θα πάμε σπίτι μας, αλλά αυτό θα υποσκάψει την αξιοπιστία μας. Παρεμβάσει των βουλευτών, το ρόλο θα πάρει η εκπρόσωπος η Έχετε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ε, κάνω κάποιες τελικέ τελικές παρατηρήσεις. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ενδιαφέρουσα ε, η συζήτηση αυτή με πολλές διαφορετικές απόψεις ε, και ήθελα να σας επενέσω για ε, το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον σας ε, και ε, την ενέργεια που καταναλώνετε για το Αφγανιστάν. Αυτό φάνηκε από τη συζήτηση σήμερα. Όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι το Αφγανιστάν είναι σημαντικό για όλους μας και για τους πολίτες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει σημαντικός παράγοντας. Στην αρχή σας ανέφερα τις προτεραιότητες και τα σχέδια για το μέλλον. Επίσης, την ισορροπία που θα πρέπει να πετύχουμε ανάμεσα στην διοχέτευση των πόρων μέσω της κυβέρνησης του Αφγανιστάν και την αναγνώριση της, ε, της προσπάθειάς μας να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Ε, συνεχίζουμε να συμμετέχουμε σε ε, σημαντικούς τομείς, σε την αστυνομία, την υγεία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, το κράτος δικαίου επίσης είναι κεντρικό θέμα. Επίσης, όλα αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται στην οικοδόμηση δυναμικού εντός των τοπικών δομών. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις ε, αφγανικές αρχές να καταπολεμήσουν ε, τον, το εμπόριο των ναρκωτικών. Επίσης ανέφερα την σημασία της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της αφγανικής κοινωνίας και στις πολιτικές δομές. Σημείωσα την ε, έκθεση του κυρίου Στίβενσον ε, σημειώνω ότι ε, το νερό και η άρδευση είναι πολύ σημαντικά σε ε, πολλές χώρες. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Αρλάκη για την έκθεσή του. Προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησης για τα σημεία κλειδιά της έκθεσης αυτής και θα ήθελα κλείνοντας να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν για τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ ε, και ε, τα τελευταία του λόγια πριν την τελευταία του εγχείρηση. Ε, αυτό δείχνει ακριβώς τι άνθρωπος ήταν και θα μου λείψει πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία είπατε εκπρόσωπη, ο κύριος Αρλάκη έχει το λόγο τώρα, ο εισηγητής για να κλείσει την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να κάνω κάμια δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, είμαι πολύ ικανοποιημένο που κανένα δεν άσκησε κριτική για τέσσερα βασικά σημεία που αναφέρει η έκθεση μια μεταρρύθμιση της ε, διεθνούς βοήθειας, ε, να εξαλειφθεί η καλλιέργεια της παπαρούνας, καλύτερα, καλύτερο συντονισμό της κατάρτισης των αστυνομικών και υποστήριξη της συνεχτικής διαδικασίας. Όλες οι παρατηρήσεις αφορούσαν άλλα θέματα, όχι αυτά τα τέσσερα. Και είμαι ικανοποιημένο που μετά από ένα χρόνο συζητήσεων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, οι συνάδελφοι επιβεβαίωσαν την υποστήριξη στη δομή τουλάχιστον, τη βασική δομή, το σκελετό της ε, έκθεσης η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτή είναι η έκθεση που με 60 ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά, ε, σχεδόν ομόφωνα δηλαδή, έχει εγκριθεί. Έχουν ενσωματωθεί διάφοροι συμβιβασμοί ε, που συμφώνησαν διάφορες πολιτικές ομάδες επίσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το πραγματικό κείμενο της έκθεσης, το τελευταίο κείμενο. Κύριε Ζουβά, θέλω να σας πω το εξής. Δεν μιλάμε πουθενά για δυνάμεις κατοχή του Αφγανιστάν. Αυτό το έλεγε το αρχικό κείμενο. Το τελικό κείμενο λέει για το συνασπισμό διεθνών δυνάμεων που είναι επιτόπου στο Αφγανιστάν. Αυτό το τμήμα της ε, έκθεσης έχει αλλάξει μέσω τροπολογίας. Ε, και το πιο σημαντικό θέμα είναι τα ανεπάνθρωτα αεροπλάνα. Αλλά όμως εγώ το αναφέρω σε δύο γραμμές, ένα συμβιβασμό. Δεν είναι μια έκθεση αυτή για αυτά τα αεροπλάνα είναι αποτέλεσμα συμβασμού των πολιτικών ομάδων. Θα μπορούσαμε να είχαμε συμφωνήσει για αυτό το θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ ε, εμπιστεύτηκα τον συμβασμό που, στον οποίο έχουμε φτάσει. Πουθενά δεν λέμε στην έκθεση ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε τα μάλα αυτά τα αεροπλάνα. Πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για το θέμα των επάνδρων αεροπλάνων. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, ευχαριστώ και την κυρία Άστον. Ελπίζω να λάβει υπόψη το περιεχόμενο της έκθεσης, ε, που είναι πολύ συγκεκριμένο και, για, και μιλάει για μια στρατηγική εξόδου από το Αφγανιστάν. Κύριε Σιγητά, ε, δέχεστε μια ερώτηση, δέχεστε κύριε Σιγητά μια ερώτηση από τον κύριο Ζεγκέντη να, ο, ο συνάδελφος ο κ. Ζαγκέντη θέλει να σας υποβάλει μια ερώτηση. Σήκωσε μπλε κάρτα. Yes. Okay. Ε, κύριε συνάδελφε, μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτησή σας στον εισηγητή. Μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Σύντομα σας παρακαλώ. Κύριε Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω την εξή ερώτηση. Δεν την απευθύνω στον κύριο Αρλάκη, αλλά σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, απευθύνω την ερώτηση. Μία προειδοποίηση, ας πούμε, ή μία ανησυχία. Εγώ είμαι μη εγγεγραμμένος και δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να συνεισφέρουμε στη συζήτηση. Ε, προσήλθα μία ώρα ε, νωρίτερα και είπα στο προσωπικό σας, στη γραμματεία, ότι θα ήθελα να μιλήσω και εγώ σήμερα. Δεν μπόρεσα και θα υποβάλω τα σχόλιά μου γραπτός, αναγκαστικά. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να δείχνετε μεγαλύτερη κατανόηση προς τους μη εγγεγραμμένους που έχουν πολύ, πολύ περιορισμένη ευκαιρία να λαμβάνουν το λόγο. Oui. Διαδικαστικό θέλετε. Να διορθώσω αυτό που υπόθηκε. Ο κύριος Σαρλάκη έχει δίκιο. Το τελικό κείμενο που μας προτείνει δεν μιλάει στο εκτιμώντας ε, β την έκφραση δυνάμεις κατοχής. Απλώς η μετάφραση, η η γαλλική μετάφραση δεν ε, ε, διορθώθηκε. Μέχρι σήμερα το πρωί η γαλλική μετάφραση μιλούσε για δυνάμεις κατοχής. Εξού και η παρέμβαση του κυρίου Ζουβά. Διαδικαστικό, κύριε Ντονζόν, αυτό. Ε, ο κύριος Ντανζόν δεν έκανε point order, δεν επενέβη για, για point order και ο κύριος Σεντέκη ε, σήκωσε την μπλε κάρτα. Προσέξτε κύριε συνάδελφοι, η μπλε κάρτα δεν αντικαθιστά το χέρι.